Good morning everybody. Dear colleagues, dear... Uh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί επισκέπτες, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε με τη δεύτερη μέρα της συνεδρίας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Καταρχήν να σας αναγγείλω μια μικρή αλλαγή. Το σημείο 16, η έκθεση Σνέλχαρτ, θα ψηφιστεί σήμερα αλλά το απόγευμα. Το σημείο 16 λέω. Υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα. Αναβάλλεται για το απόγευμα η ψηφοφορία της έκθεσης Νέλχαρτ. Έχετε λάβει και την τελευταία πρόταση Κράμερ και Βάις Γκέρμπερ μετά τη χθεσινή συζήτηση. Θα την ψηφίσουμε μετά το σημείο 17. Ε, θα έχουμε το επίμαχο σημείο για τους λαμπτήρες και την ε, επιτροπολογία. Έχουμε και μία πολυμελή ομάδα επισκεπτών ε, της κυρίας Ντάγμα Ροτμπέρεντ, ψηφοφόρων της κυρίας Μπέρεντ. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε συνεδρίαση μας στη διάρκεια της ημέρας, Ιδιαίτερα συζήτηση για τους ε, λαμπτήρες φωτισμού. Ε, ίσως μας επισκεφθεί και κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο από τη Γερμανία. Α, δεν θέλετε. Καλά. Θα ψηφίσουμε αν θα δεχτούμε το τηλεοπτικό συνεργείο ή όχι. Έχουμε και ένα κατακένουργο μέλος στην ε, στη γραμματεία, τη Μάρτσελα Γκράζελ. Την καλωσορίζουμε. Η Μάρτζελα Γκράζελ ε, είναι στη γραμματεία και κατάγεται από την Τσεχία. Παρακαλώ, μπορείτε να σηκώσετε, Μάρτσα να σας δουν οι συνάδελφοι. Τελευταία ανακοίνωση. Σας έχουν μοιραστεί δοσιαί για τη λωρίδα της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τον Υπουργό Υγείας της Αιγύπτου που ζήτησε την υποστήριξή μας για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Του υποσχέθηκα λοιπόν να σας μοιράσω όλες τις πληροφορίες που μου έδωσε ο Αιγύπτιος Υπουργός Υγείας. Εξού και τον ντοσιέ που έχετε λάβει με στοιχεία για τη λωρίδα της Γάζας. Σημείο 10 τώρα στην ημερήσια διάταξη προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Έκθεση της Φρεντερίκ Ρίς. Ερωτώ τη Φρεντερίκ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας την ψηφοφορία ή έχετε να προσθέσετε κάτι κυρία Ρίς. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε μόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για το ζωηρό ενδιαφέρον που έδειξαν για την έκθεση και τις πολυάριθμες τροπολογίες που κατέθεσαν. Παρόλο που δεν θα τις υποστηρίξω όλες, προσπάθησα να διασφαλίσω μια ισορροπία στην έκθεση μεταξύ της προστασίας της υγείας των ε, Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά ε, και της επικουρικότητας για τις ε, τροπολογίες παραγράφου 1 που είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλούν για πιο απαιτητικά όρια έκθεσης για το σημείο αυτό μιλήσαμε στην Ολομέλη σε προηγούμενη μας έκθεση για το περιβάλλον και την υγεία το Σεπτέμβριο του 2008. Μαζί με τον καθηγητή Τρακατέλη και την κυρία Φερέιρα είχαμε υποβάλει τη σχετική πρόταση και είχαμε υποστηριχθεί από την Ολομέλεια σύσσωμη σχεδόν. Τώρα, η τροπολογίες 14 και 15 Βανίστερο και Μπέργκερ ουσιαστικά επαναφέρω ένα θέμα που έχει ούτως ή άλλως γίνει ομόφωνα δεκτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να το επαναφέρουμε για να είμαστε συνεπείς με προηγούμενες μας εργασίες. Ό,τι αφορά αυτά τα όρια έκθεσης, 41 βολτ το μέτρο είναι το όριο στην Ευρώπη, ενώ 8-9 χώρες, ή περιφέρειες είναι πιο απαιτητικοί και αυστηροί στις προδιαγραφές τους. Η περιοχή της, ε, των Βρυξελών θα περάσει στα 3 βολτομέτρα στις 15 Μαρτίου, ε, ανησυχώντας και για την υγεία των Ευρωβουλευτών, γιατί στην εμβέλεια αυτής της περιφέρειας βρίσκεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς καμία συνέπεια ή δυσκολία σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις και την πρόσβαση στα δίκτυα. Από τις 15 Μαρτίου λοιπόν ισχύουν και στις Βρυξέλλες αυστηρότερα όρια έκθεση, 3 βολτ το μέτρο. Σας ευχαριστώ. Θέλει άλλο κανείς από τους σκιώδεις ηγητές το λόγο ή μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ετοιμάστε τους καταλόγους ψηφοφορίας παρακαλώ και τις ε, κάρτες τις ηλεκτρονικές. Μια στιγμή ζήτησε το λόγο η κυρία Αγιάλα. Μία προειδοποίηση μόνο, γιατί δεν υπάρχει στον κατάλογο. Η προφορική τροπολογία 27 της κυρίας Μπέργκερ έχει προσθέσει την τελική παράγραφο «Καλή την βιομηχανία και τις αρχές. Και τις αρχές. Ένα λάθος ε, τυπογραφικό έγινε εκεί, έλειψε, παραλήφθηκε το και. Και τις αρχές λοιπόν προστίθεται. Καλώς, εγώ έπρεπε να το είχα αναγγείλει. Σας ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε κυρία Γιάλα. Αρχίζουμε λοιπόν με, τις τροπολογίες, ε, με την τροπολογία 14 και η συγκητρία είναι κατά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 14 του κ. Βανίστερο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 19 υπέρ 21 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Τέλος. 25 υπέρ, 19 κατά. Δίκιο είχατε, εγκρίνεται η τροπολογία 13. Next Η επόμενη καταπίπτει, τροπολογία 16 της Σύνοτ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ποιος είναι υπέρ Αδάμου και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, η 17 καταπίπτει, οπότε περνάμε στη 18, Λούκας Ισλερμπεγιά Αδάμου, κατά τμήματα ψηφοφορία, υπέρ του πρώτου τμήματος, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 18 δεύτερο τμήμα. Τέλος. Ψήφισαν 32 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ, σύνοτ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20, σύνοτ, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 20. The vote closed. Τέλος ψηφοφορίας, 33 υπέρ, 10 κατά, σαφώς εγκρίνεται. 21, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, τροπολογία Κατά τμήματα ψηφίζουμε. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογή 24. Αγιάλα Σέντερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 15 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. 27 προφορική τροπολογία. Έχετε λάβει την μικρή διόρθωση. Ποιος είναι υπέρ της 27. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Καλά, ηλεκτρονικός έλεγχος αν θέλετε, για την 27 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 12 υπέρ, 32 κατά. Σαφώς απορρίπτεται. 28 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Να την ψηφίσουμε. 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει 36, Πέτερλε, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 σύνοτι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 39 κατά τμήματα ψηφοφορία, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40, ποιος είναι υπέρ, κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 40. Αδάμου, Λούκα και Μπεγκά. Τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ 41, Αγιάλα Σέντερ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, απορρίπτεται. 43, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46, υπέρ. Κατά, Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 46. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Ισοπαλία 23 υπέρ 23 κατά. Απορρίπτεται. 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ κατά εποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 22 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 5 της κυρίας Σύνοτα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ψήφισαν 32 υπέρ και 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Amendment. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 37 υπέρ και 10 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Who against? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Να πάρω. 43 υπέρ, 3 αποχές, μια ψήφος κατά, με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίθηκε η έκθεση. Χαρητήρια θερμά κυρία Φρεντερίκ Ρίς. Okay, Mr. a point of order. Ο κ. Ε, Μουσάκης, ένα ε, διαδικαστικό θέμα, παρακαλώ. Chiedo scusa, eh, volevo avere... Συγγνώμη, θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δυνατόν κύριε Πρόεδρε να ψηφίσουμε τη δική μου έκθεση για την αλία. Γιατί μια αντιπροσωπεία ασθενών, ε, ψυχικά ασθενών που έχουν φτάσει χρειάζονται με χρειάζονται για να μπουν στο κτίριο. Είναι πολύ σύντομο. Παρακαλώ συνάδελφοι, αν γίνεται να ψηφίσουμε τώρα τη δική μου έκθεση. Sono pochissimi voti, quindi... Είναι ελάχιστες ψηφοφορίες. Item okay. Are there here any objections for, for changing agenda? Έχει κανείς αντίρρηση αυτό, όχι συμφωνούν όλοι. Κράμε διαδικαστικό. Ένα δευτερόλεπτο. Ήθελα να πω ότι κανονικά δεν λαμβάνουμε υπόψη τέτοια προσωπικά προβλήματα και ραντεβού. Λοιπόν, εάν διαφωνεί κάποιος δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Okay, so exceptional... Λοιπόν, κάθε εξαίρεση, κάθε εξαίρεση. Ποιο είναι το θέμα σας ακριβώς, το 18. Ωραία. Σημείο 18, έκθεση του κύριου Μουζάκιο. Προετοιμαστείτε για την ψηφοφορία του θέματος αυτού. Ελπίζω ο να μην θέλει το λόγο. Ωραία. Ψηφίζουμε τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Τροπολογία 4, παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος, η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 35 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Δύο ταυτόσημες, οι 8 και 9, υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορία. 22 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτονται. Η επόμενη καταπίπτει. Η 5 παρακαλώ του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, Ένα τροπολογία ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία The vote is closed. Πέραση τη ψηφοφορία. 45 υπέρ, 2 κατά, 1 αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μουτσάκιο. Okay, colleagues, don't laugh. Elections are coming, so... Ε, ε, Λοιπόν. λοιπόν, το επόμενο σημείο είναι το σημείο 11, έκθεση της κυρίας Καρολάιν Λούκας. Θα ήθελα να τη ρωτήσω αν μπορούμε μέσα να περάσουμε ψηφοφορία. Ναι, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. So, let me start with compromise. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 4 ενωμένη 4 τροπολογία We are checking compromise, compromise consolidated 4. Ενωπημένη 4 λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 και 16 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές για να ελέγξουμε. Ενοποιημένη 18. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. Everybody has Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 35 υπέρ, 9 κατά, μία αποχή, ενεκρίθη. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 22 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε. 22. The vote is closed. Πέρας 36 υπέρ, 11 κατά, καμία αποχή. Ένα κρύφη. Ενωπημένη 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενωπημένη 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν για να δούμε τώρα περνάμε στο πολυγιά 12 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκατρία, ωραία. Δεκατρία, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. δύο. υπέρ. Κατά αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άχρη ψηφοφορία. Την 102 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέραση ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 12 κατά. κρίθη. Δεκατέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάμε στην 19 της συζητήτριας υπέρ. Ακούγονται φωνές 17. Α, ναι, ναι, την παρέβλεψα αυτή. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. 17, 17. Της κυρίας Λούκας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 18. Υπέρ. Α, όχι 18, 19, 19. 19. Συγγνώμη. Η 19 της κυρίας Λούκας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν έχω πάρει μπρος ακόμα. Σε μία ώρα τόσα λάθη έκανα. Η επόμενη καταπίπτει, έχει αποσυρθεί, αποσυρθεί. 24. Έτσι, σωστά. 24. Ποιος είναι υπέρ της 24. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Twenty-five. Okay, amendment 25, who in favor. Λοιπόν, 25, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Now let me put the vote on the button. 8. Για να δούμε. Είναι τα 8 υπέρ. Στην ίδια σελίδα κάτω-κάτω είναι στο δικό μου τη λίστα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139. Για να δούμε. 140. τάχα, Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραβλέψαμε το 139. Ποιος είναι υπέρ. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 σελίδα 151 τροπολογία. 151. Υπέρ. Ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία. Δεν βλέπω ότι πρέπει να έχει καταπέσει. 151 λοιπόν. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. If I'm right, Αν δεν κάνω λάθος, άρθρο 6, τροπολογία 34 είναι αυτή που θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Διαδικαστικό, με συγχωρείτε. Δεν το είχα δει αυτό. Η 151 θα πρέπει να έχει καταπέσει νομίζω. Γιατί για δείτε τι λέει στην, το κάτω-κάτω τμήμα της προηγούμενης σελίδας. Ε, είναι μαζί με τις άλλες, δηλαδή 148, 149, 150 και 151 αναφέρονται στο ίδιο σημείο και πάνε μαζί. Και έχουν καταπέσει επειδή υιοθετήθηκε η συμβιβαστική 16. Okay, I'm... Α, ναι. Εγώ δεν είχα την ένδειξη αυτή, αλλά πραγματικά ανήκει στην επόμενη σε ομάδα. Για την 151 ε, μιλήσατε, έτσι. Ωραία, την ψηφίσαμε, αλλά εντάξει, έχει καταπέσει, δεν έχει, δεν έχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, επιτρέψτε μου να περάσω στην Τροπολογία 34 για το άρθρο 6 της συζυγήτριας. Είναι σωστό? Η 158 νομίζω. Την παραβλέψατε κύριε Πρόεδρε. 158. Που λέει ότι είμαι συμβατή. Ή όχι. Άρθρο 5 παράγραφος 1. Yeah. Okay. If my file is right, there is written that Εάν έχει δίκιο το κείμενο, έχουμε εδώ δύο τροπολογίες, 100 με 7 και 100 με 8 και λέει ότι ε, καταπίπτουν εάν υιοθετηθεί η συμβαστική 16. Έτσι δεν είναι. Ωραία, η συγκέντρια συμφωνεί. Ωραία. Λοιπόν, 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 10. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 46 υπέρ. Κανένα κατά. Όλοι ψήφισαν υπέρ λοιπόν. Δεν φαινόταν έτσι με την ανάταση χειρός καθόλου. Νομίζω τα μάτια μου δεν έχουν πρόβλημα. Εσείς αλλάζετε την άποψή σας. Α, μήπως είναι ο φωτισμός κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Καλώς. Λοιπόν, για να κοιτάξουμε τώρα. 187. Ωραία. 187 λιωτάχ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται δύο γλωσσικές, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Η 43 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 188 κρούπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 188. 188. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 21 κατά. Ενεκρίθη. Είναι τα 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Κρούπα 189. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Η 190 υπέρ κατά για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 190 παρακαλώ πέρασε της ψηφοφορία. 25 υπέρ 21 κατά εκρήθη 192 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. 198 και 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201. Εκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 Λούκας υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας 36 υπέρ 13 κατά ενεκρίθη ξεκάθαρα 203 ο Κόρχολα Ματιού, υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο να ψηφίσουμε όταν έχει τόση φασαρία στην αίθουσα. Στην επόμενη σελίδα. Τροπολογία 47. Κρούπα. Υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. Leotard, who is in favor? Who is against? 48 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, Λούκα υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 49, εκ υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 51 με μια προφορική τροπολογία των πρασίνων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. 56 κρούπα. Ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. The vote is closed. Πέρασε 26 υπέρ και 25 κατά. Ενεκρίθη. 58. Μούλαρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 λούκα υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. Ίντα 1 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 59 κρούπα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 63 λιωτάρ Everybody has voted. The vote is closed. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφορές. 32 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή. Ενεκρίθη. Είναι τα 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη είχε υποσύρθει. Η επόμενη καταπίπτει. 66 υπέρ. Κατά αποχές. Για να ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά Είναι 66. The vote is closed. 35. υπέρ, 15 κατά. κρίθη. 68. Λούκας υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω κανένα χέρι να σηκώνεται. Για να ελέγξουμε. 68 Λούκας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. 36 υπέρ 18 κατά. εκρήθη. Εβδομήντα. Γιωτάρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε αν θέλετε για την 70 λιωτά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 22 κατά. Δεν εκρήθη. Τρεις, τέσσερις ταυτόχρονες. 7, 71, 72 και τα 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελευταία σελίδα η 77 εκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο ταυτόχρονα 8 και 79 Α, όχι, καταπίπτων, συγγνώμη. Η 80, κορφόλα ματιού, υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 80, κορφόλα ματιού. Πέρας πληροφορίες. 19 υπέρ, 33 κατά. Α, περίφθη. 81 λιωτάρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η επόμενη, για να δούμε, για την 82. Καταπίπτει. 83. Κρούπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 87 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας ψηφοφορίας 27 υπέρ 26 κατά ενεκρίθη συγχαρητήρια 88. Εκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη. 89. Εκ με μια προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Κρούπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. πέρας ψηφοφορίε. 54 υπέρ, μία ψήφο κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Λούκα. Thank you. Yeah, Thank you very much indeed. Thank you. Next item on our agenda is uh, item 12, which is... Uh, Περνάμε στο σημείο 12, που είναι η ψηφοφορία για την έκθεση της Λίντα Μακάβαν, δηλαδή η κούση συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Το είμαστε. να ρωτήσω την εισηγήτρια αν μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, προετοιμάστε λοιπόν τους καταλόγους ψηφοφορίας σας, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Να περιμένω μερικά δευτερόλεπτα ώστε να μοιραστεί ο κατάλογος ψηφοφορίας. Όλοι έτοιμοι. Ωραία λοιπόν. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 46 καταπίπτει. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Παίρνουμε την τροπολογία 12. Ε, ψηφίζουμε μάλλον την τροπολογία 12. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 19 κατά, εκρίνεται. <clears throat> Τροπολογία 13 υπέρ, κατά. Τέσσερα χέρια είδα μόνο να σηκώνονται. Λοιπόν, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Οι δύο, οι επόμενες δύο καταπίπτουν. 54 βάζει Γκέρμπερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 χόλμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 14 Τέλος ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 29 κατά απορρίφθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 17 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 χόλμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16, 60 ε, ε, μάλλον πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 19 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. Τροπολογία 61. Α, καταπίπτει. Και η επόμενη. Ωραία, προχωράμε στην 19 στο δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60, τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 60, τρίτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. 19 τρίτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 19 τρίτο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 62 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22ο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν 64 σαρτόρι υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 62 τέταρτο τμήμα υπέρ να ελέγξουμε, να ελέγξουμε τη σαρτόρι 64 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 64. Τέλος της ψηφοφορίας. Όχι. Αδύνατον. Όχι, δεν είναι δικό μου λάθος. Όχι, δεν σηκώσετε τα χέρια σας. Εντάξει, εγκρίνεται. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία κιόλα. Ε, ε, τροπολογία 23ο ε, τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 62 πέμπτο τμήμα. Υπέρ. κά καταπίπτει. Δύο ταυτόσημες. 62 έκτο τμήμα και 63 τρίτο τμήμα. <laughs> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 63 <clears throat> τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Μάλλον. Η επόμενη καταπίπτει. Άντε την 63, αλλά έχετε δίκιο, εγκρίνεται. 63 τέταρτο τμήμα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της πληροφορίας 39 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει 65. Σαρτόρι υπέρ κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται για την 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 σερτόρι υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά 66 Τέλος της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται, 67 υπέρ. Κατά. Ελέγχω ηλεκτρονικά για την 67. Τέλος ψηφοφορίας. 41 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται σαφώς. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, 70 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά να το ελέγξουμε 74 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τέλος υποφορίας 21 υπέρ 33 κατά απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές ε, ε, εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά 78 τέλος ψηφοφορίας 20 υπέρ 23 κατά απορρίπτεται 79 χωριστή ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 σαρτόρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 ταυτόσιμες 85-86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 88. Ζίμπερ Μπέργκερ. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. 21 υπέρ 32 κατά. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 ε, χωρίς ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο, ε, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, με συγγνώμη, αλλάξουμε ηλεκτρονικά για την 97. 97 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ. 26 κατά απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99. Με προφορική τροπολογία, διαδικαστικό. Εμείς είμαστε κατά της ε, προφορικής τροπολογίας. Εντάξει λοιπόν. Άρα λοιπόν πρέπει να το ψηφίσουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. Ωραία λοιπόν. Υπέρ της 99. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευρύνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται. 102 χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 102. Τέλος ψηφοφορίας. 27, 27. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και αυτο ελεκτρονικη Ηλεκτρονική ψηφοφορία, τρίτο τμήμα. Τέλος ψηφοφορίας. 27-26. Εγκρίνεται. 31 καταπίπτει. Ε, δεν ξέρω αν το τρίτο τμήμα έχει νόημα από μόνο του. Δεν είμαι βέβαιος. Αλλά υπερψηφίστηκε έτσι. Μετά θα πρέπει να το ελέγξουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα αν έχει νόημα. Να ψηφίσουμε την 31. Υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα παρατήματα. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη έχει καταπέσει επόμενες και περνάμε στην τελευταία σελίδα. 112, δώδεκα, ναι. Ψηφίζουμε. 112. δώδεκα. Υπέρ κατά. Αποχές. Να ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 113 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Δύο. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ κατά. Αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτει. 44 χόλμα υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε τη 44. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 και 3 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σχέδιο έκθεση όπω τοποποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. 52 υπέρ, ένα κατά μια αποχή. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, επίσης ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορία 52 υπέρ, 1 κατά, μια αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Μακάβαν, την συγγήτρια. Okay. Next item on our agenda is item 13. Report Περνάμε στο επόμενο σημείο, στην έκθεση 13 του κυρίου Σαλβατόρε Ταταρέλα. Κύριε Σιγητάν, πώς θα μπορούσαμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Yeah. Thank you. Grazie. So, uh, let me start The voting procedure with... Uh, Άρχεται η ψηφοφορία της έκθεσης Ταταρέλα με δύο συμβεστικές ε, τροπολογίες που θα ψηφιστούν από κοινού. Τροπολογίες 1 και 6. Ποιος είναι υπέρ των δύο συμβαστικών τροπολογιών. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε ποιες τροπολογίες καταπίπτουν. Πολλές. Πάμε κατευθείαν στην επόμενη σελίδα. 53. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 53 συμβαστική 5 ποιος είναι υπέρ ε, μάλλον ήτρα 13 ποιος είναι υπέρ ηλεκτρονικά καλύτερα για την ε, τροπολογία 13 της ήτρα άρχεται ψηφοφορία Τέλος. Ψήφισε. 38 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 τεμπλάσιο υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία για την 54 τέλος 35 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται Η 6 καταπίπτει. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 57. Οι άλλες δύο έχουν καταπέσει. Τροπολογία 58. Προφορική τροπολογία Greens. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Bowies κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η οκτώ καταπίπτει. Ήτρε 14, Ποιο είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 ε, 61. Κορμπέι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 29 against. 19 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται. Number 9. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η επόμενη καταπίπτει. Ήτρα 16 κατευθείαν. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. 28. Τέλος ψηφοφορίας. 28 υπέρ 21 ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ήτρε 17 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. Περνάμε στην 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία η επόμενη καταπίπτει. Οι δύο επόμενες 71 και 15 και η 19 και πολλές άλλες. 57 του John Boy. Ποιος είναι υπέρ. 77 συγγνώμη. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 76. Τέλος. Ψήφισαν 32 υπέρ και 19 κατά, έχει σαφώς υπερψηφιστεί. Η 76, οι επόμενες καταπίπτουν. 77 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 77 λεπέχ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 37 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 79 σε υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 17. The vote is closed. 19 in favor, 34 against. It has been rejected. 78 uh, Sartori Bowis. Who is in... Απορρίπτω το δεύτερο τμήμα της 17, 78 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 78, Σαρτόρι και Μπόις. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 29 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν, τροπολογία 18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά, αποχές, Ούτε ένα χέρι δεν σηκώνουν οι σοσιαλιστές. Ποια είναι η θέση των σοσιαλιστών. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 81. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 8 υπέρ, 41 κατά. Απορρίπτεται σαφώς, σαφέστατα. Ήτρε. Ήτρε 25. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 82. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 33 υπέρ 17 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 83 καταπίπτει. Η 326. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Ήτρε 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 33 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Οι επόμενες τέσσερις καταπίπτουν. 85 δεν μπλάζει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 22 καταπίπτει. Η 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο πανομοιότυπες, Η 28 ή 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ήτρε 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 is in favor. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία Ήτρε 33. Άρχεται. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας 38 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 24 του συγκεκριτού. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μκο 13 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΙΜΚΟ 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται ΙΜΚΟ 13. 88 δεν πλάζει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89. Χάσει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90. Δεμπλάζιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91. Δεμπλάζιο. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 91 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, 30 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Η επόμενη καταβίωτη, 26, 27 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 28, ποιος είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Η επόμενη, η ΜΚΟ 14 καταπίπτει. 95 Ο Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 95. Οι προηγούμενες έχουν καταπέσει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 95. Τέλος. 48 υπέρ. 5 κατά. Χωρίς αποχές. Σαφώς εγκρίνεται. Η τροπολογία 95. 102 τώρα. Λέμπεχ, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 ήτρε, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 γκαρντίνι, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 35, ΙΜΚΟ 15, πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, την Ήτρε 35 και την ΙΜΚΟ 15, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, 34 υπέρ 20 κατά, εγκρίνονται. Τροπολογία 104, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Οι επόμενε 2, 30 και 31 καταπίπτουν. 32 Λέμπεκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 32 Λεμπεκ. Ποιο ειναι υπερ κατα Αποχέ. ηλεκτρονικος ελεγχος για την τροπολογια 32 λεμπεκ αρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ψήφισαν 38 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Ή 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 33. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 30 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ. Τριάντα τέσσερα. Υπέρ. Μα δική σας είναι η πρόταση. Όχι όμως και της ομάδας. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Ήμκο 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την Ήμκο 1. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος 35 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. 36 Σαρτόρι. Ποιος είναι υπέρ. Σαρτόρι Μπόουις. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικό έλεγχο τροπολογία 36, Σαρτόρι και Μπόουις. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 25 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά, οχές, απορρίπτεται. Ήμκο 2, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μάλλον έχει απορριφθεί αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά για ασφάλεια ΙΜΚΟ 2 άρχεται η ψηφοφορία Vote is closed now. 25 in favor, 27. 25 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. 37 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 38. The vote is closed. 42 Τέλος ψηφοφορίας, 42 υπέρ, 11 κατά, με εμφανή διαφορά εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει, η 40. Ήτρε 4, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Ή μάλλον ε, έχει καταπέσει. 41. Ποιος είναι υπέρ. Βέικμεν Ντόιλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η Ήτρε 5 και η 3 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικός έλεγχος για τις ΙΤΡΕ 5 και ΙΜΚΟ 3. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 30 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Ήτρε 6. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 43. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 42 καταπίπτει. Ήμκο 4. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Η 37. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Η 38. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 45 καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed 52 52 υπέρ, μία ψήφος κατά και δύο αποχές. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχιδη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 51 ψήφισαν υπέρ, κανείς κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σαλβατόρε Ταταρέλα. Θερμά συγχαρητήρια. Var det var John? in the, in the, um, Πρόεδρε, στο κατάλογο ψηφοφορία για το κείμενο που ψηφίσαμε όλοι τώρα υπάρχουν κάποιε υποσημειώσεις στα Ιταλικά. Τα Ιταλικά μου δεν είναι τόσο καταπληκτικά, αλλά εκείνη για την 82 λέει κάτι κόστη αλλά σπέζε. Αυτό σημαίνει ότι ελπίζουμε να έχουμε καφέ. Okay. Yeah, there is, there is proposal for... Υπάρχει πρόταση για καφέ. Ωραία. Να το οργανώσουμε. Συμφωνεί. So, next item. Επόμενο θέμα. So there is one, one announcement before we start, uh, start... Μια ανακοίνωση πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Υπάρχει μια πολύ πιο πρόσφατη εκδοχή του γράφου αυτού και ίσως ορισμένοι δεν το έχουν. Με μια μικρή αλλαγή μόνο για την τροπολογία 72. Φάση. Για το άρθρο 16 σημείο 1 υποπαράγραφος 1 Ένα σημαντικό τμήμα της υποπαραγράφου παραμένει, το 1α όμως έχει κάπως μετατεθεί. Πριν από την 73. <clears throat> το σας το λέω από τώρα. Δηλαδή για το άρθρο 16 παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α νέο. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσίβη που είναι η εισηγήτρια να μπορούμε αμέσως να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θα προτιμούσα βέβαια να ξεκουραστώ λιγάκι, αλλά δεν μου δίνεται δυνατότητα. Καλύτερα να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Θα ήθελα να αρχίσω με την τροπολογική παριθμών 9. Κράμερ Βάις Κέρμερ. Για να, απορριφθεί το, σύνολο της πρώτης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 24 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρα 13 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Σαφώ δεν εκρήθη. Τροπολογία 40 φοβλέτα υπέρ, κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα δύο υπέρ. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι τρεις επόμενες καταπίπτουν. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η... η επόμενη, η επόμενη, 50, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 και 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Οι δύο υπόλοιπες καταπίπτουν. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρα 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 67 παρακαλώ. Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 43 υπέρ 12 κατά. Ναι, ναι, ναι. Ενεκρίθη. Η επόμενη καταπίπτει. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οι επόμενες δύο καταπίπτουν. 18 ήτρε το ενολόγο σημείο υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 7. τα εν λόγω σημεία του της 7. Ψηφίσουμε. Yeah. Okay. I put it to the Ωραία, ψηφίσουμε. 72, το λόγω. 7 τα εν λόγω σημεία υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 και ήτρε 19 ταυτόσημες υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 75 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ιτολικέ σκέψει. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δύο τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 24. Πέρασε ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 5 κατά διαφορετική κατάσταση από αυτή που είχα δει. Ήτρε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. 27 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η χρονική σκέψη 23, δύο ταυτόσημες τροπολογίες 38 και ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ήτρε 10 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ήτρε 10 Άρχιψη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 24 υπέρ, 30 κατά, περίφθη. Ή 30 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε και αυτό. Ή 30. Πέρυσι φορά 41 υπέρ, 14 κατά. κρίθη. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο της τροποποιημένης έκθεσης ηλεκτρονικά παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ε, ε επίσης ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά επίσης. The vote is closed. οι 46 υπέρ, 5 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια. Μουτσίβη.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 So, my dear colleagues, I understand that, that you are very tired, yeah. as I am, but let me... Λοιπόν, ε, βλέπουμε τι θα γίνει με το καφέ, αλλά περάσουμε στο σημείο 15 για την εμπορία διοκτώνων προϊόντων η έκθεση Ντασιάν Οκτάβια Σάρμπου. If it's possible to vote on block. Μπορούμε να ψηφίσουμε ο μπλοκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μία εξαίρεση. That, uh, only and Οι τροπολογίες 7 και 4 θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. Το σύνολο της τροποποιημένης ε, έκθεσης ε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχιε ψηφοφορία τώρα. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίες. in favor, no one against, no abstention. 52 υπέρ, κανένας κατά, καμία αποχή. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ηλεκτρονικά No. Okay. I'm waiting, waiting, because I see that no one, so so many members doesn't vote. Now the vote is closed. Λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορίες. 51 ψήφοι είπε. κανένας κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Σέρβου. So, uh, because uh, as we decided uh, that... Uh... Αποφασίσαμε ότι η έκταση Σνέλχαρ θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην έκθεση Παλέτκη. Γκίτο, έχει το λόγο. Μια πολύ σύντομη ανακοίνωση, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά υπήρξε ένα λάθος στην ε, λίστα, στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, στην 222 λοιπόν η, ψηφο... η ψήφος μας είναι θετική. Αυτό για τον κατάλογο ψηφοφορίας των σοσιαλιστών. Για να μην διακόψω την ψηφοφορία. Ναι. Μόνο λοιπόν για να ενημερώσω το... τα μέλη. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. If I understand it's information for the socialist group. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα αυτή η ενημέρωση αφορά τους σοσιαλιστές. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα λαθάκι στον κατάλογο της ψηφοφορίας σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, τον κύριο Παλέτσκι. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με την τροπολογία 69 σε δύο τμήματα. Το σνίπερ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. The vote is closed. 27 in favor, 20 against. It has been carried. The second part. Εγκρίνεται 27 προς 20. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε επίση. The vote is closed. Πέρασε 30 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται επίση. 68. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρει ταυτόσημε. 71, 72, 73. Υπέρ. Α, κατέπεσαν όμως. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε την 74 λιωτά ηλεκτρονικά. The vote is closed. Τέλος 18 υπέρ 29 κατά. Ναι, ναι. Απερίφθη. 77. Πράιερ. Με μια προφορική τροπολογία. Υπέρ. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό της υποβάλλουσας. Είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας, Πρόεδρε. Ωραία. Ψηφίζουμε χωρίς την προφορική τροπολογία, λοιπόν. 77 χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76. Φερέρα με μία προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. me check it by electronic vote, but there is... Ηλεκτρονικό σας διαδικαστικό θέλετε. Είμαι κατά και αυτής της προφορικής τροπολογίας, Πρόεδρε. Okay, so, so, yeah. There is objection to oral amendment. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφωνία για την προφορική τροπολογία. Και για την τρίτη περίπτωση πάλι διαμαρτύρεστε. Ναι. Να μας το πείτε από πριν άμα είναι. Γιατί κατά διάρκεια διαδικασία είναι πολύ πιο δύσκολο. Λοιπόν, και οι τρεις τροπολογίες χωρίς την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, 76 χωρίς, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 75 χωρίς προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά, για να το ελέγξουμε αυτό. 75. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 25 κατά. Να περίφθει. 78, Ντόιλ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. 78. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 30 κατά. Απερίφθη. 79 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 81. Να ελέγξουμε την 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας πληροφορίας 26 υπέρ, 24 κατά. Είναι κρίθη. Σας ευχαριστώ. 81 Φεραίρα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Νομίζω ότι απερίφθη. είναι να το ελέγξουμε όμω ηλεκτρονικά. Για την 81. The vote is closed. Πέρασε στις 14 υπέρ, 33 κατά. Απερίφθη σαφέστατα. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω κανένα σηκώνει τα χέρια του. Για να ελέγξουμε την 80. Πέρασε ψηφοφορίας. 57 υπέρ. 9 κατά. Εγκρίνεται σαφέστατα. 4 ταυτός όμω. 85, 83, 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. ψηφοφορία. 22 υπέρ, 26 κατά. Απερίφθησαν. Τα επόμενα τρία ταυτόσημα. 86, 87, 88. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φορέ 35 υπέρ, 15 κατά. Ενεκρίθη σαφέστατα. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3 αυτόφημες. 90, 91, 92. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απερίφθη. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Θα το ελέγξω, ναι, ναι, ναι, ναι δεν είμαι σίγουρος. Άχι πληροφορία. Πέρασε πληροφορίες. 24 υπέρ, 26 κατά. Πράγματι απερίφθη. Είναι 94. Α, ήταν, πήγαινε με, με, με, τα άλλα, ναι. Πήγαινε με τα άλλα και αυτό. Μάλιστα. Απερίφθη λοιπόν. 93. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε 93, παρακαλώ. Άρχισε η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 23 υπέρ, 30 κατά. Απερίφθη. 96 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτωται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100, 101, 102, 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αυτές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. αυτές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 105. Πέρες ψηφορές. 30 υπέρ, 22 κατά. Ναι, είναι κρύφη. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν. 107 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 110, 111, 112, 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτει. 115. Μπράιερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 115. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίες. 38 υπέρ, 17 κατά. Ανακρίθηκε ξεκάθαρα. 116 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 117 Ρενά Σόμερ υπέρ. Κατά. εποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 118. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας πληροφορία 26 υπέρ 22 κατά. Ενεκρίθη. Τρεις ταυτόσημε. 119, 120, 121 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. πάμε επόμενη καταπέπτει. 122 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε. Την 122 ηλεκτρονικά. τη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 30 κατά. Απερίφθη. 131 υπέρ. Κατά. Ανεκρίθη. Next two falls. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν και οι μεθεπόμενοι επίσης. 125 Φερέρα σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά πέρας πληροφορίας 19 υπέρ και 36 κατά απεριφθεί 126 υπέρ κατά να ελέγξουμε άρχισε φορεία. πέρασε πληροφορίες 20 υπέρ 32 κατά απέριφθη 127 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 128 και 129 <clears throat> ταυτόσημες Ποιοι είναι υπέρ κάτα απόχες εγκρίνονται Α, όχι ας ελέγξουμε 128 και 129 Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 21 κατά εγκρίνονται. Τρεις ταυτόσημες, 132, 133, 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 136 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 136. Τέλος ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες, 139, 140, 141, υπέρ, κατά αποχές το ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. Τρεις ταυτόσιμες. 143, 44, 45 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. 25-35 κατά απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ Κατά. Να ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. 149 υπέρ. Ε, συγγνώμη, έρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. 17... Τέλος ψηφοφορίας, 17 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152. Φέλνερ με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 153. Τέλος ψηφοφορίας. 37 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 154. The vote is closed. 30 in favor, Τέλος ψηφοφορίας, 30 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες, 155, 56, 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Επόμενη ψηφίζουμε την 158 Φιέλνερ. Ρενάτε Σόμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 χωριστή ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 24 κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται επόμενη καταπίπτη 165 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά Τέλος ψηφοφορία 19 υπέρ, 35 κατά απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Απογές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες. 171 και 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 173 Α, θέλετε να αλλάξουμε τις δυο ταυτόσημες, εντάξει. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τις 171 και 172. Τέλος ψηφοφορίας, 31 υπέρ, 25 κατά, είχατε δίκιο. Έχετε δίκιο, εγκρίνονται. 173 καταπίπτει λοιπόν τότε και έχουμε δύο ταυτόσιμες 174 και 175 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά Τέλος, ε, άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας 21 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται 176 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενες δύο καταπίπτουν. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορριπτόται. Οι δύο επόμενε καταπίπτουν. 183 υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει, να ελέγξουμε. Είναι η 187 της Ρενάτε Σόμερ. Ελέγχουμε, ελέγχουμε την 187. Τέλος της ψηφοφορίας. Είχα δίκιο. 188 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 194 Τέλος ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 38 κατά απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την 195 ψηφίζουμε τέλος πληροφορίας. 34 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Είναι 196 και 197. Η... Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Τέλος πληροφορίας, 36 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Οι ε, 200 υπέρ. Κατά. Vote is closed. That is free. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 33 υπέρ 24 κατά. Εγκρίνεται. False. Η επόμενη καταπίπτει. 202. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρεις ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Τις 204, 5 και 6. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτει και δύο ταυτόσημες 211-212. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 211 και 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ah, Τώρα ψηφίζουν περισσότεροι σοσιαλιστές από ό,τι δικαιούνται. Ένας επιπλέον, ένας θα πρέπει να ψηφίζει. Ωραία. Ισοψηφία με 28 ψήφους. Απορρίπτονται. 209 Ρενάτε Σόμερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 210 Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 210. The vote is closed. Τέλος. 30 υπέρ 27 κατά. Εγκρίνεται. Η 213 κατά πίπτη. 208. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 214 και 215 ταυτόσημες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 2.14 και 2.15 και 2.16 λέει ο πρόεδρος. 2.14, 2.15, yeah. Ή μάλλον για τις 2.14 και 2.15. Ηλεκτρονικός έλεγχος, τέλος ψηφοφορίας, 18 υπέρ 38 κατά, απορρίπτονται. Άλλες τρεις πανομοιότυπες, 216, 17 και 18, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις τροπολογίες. It's check, it's check of three identical amendments. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες 216, 17 και 18. Τέλος ψηφοφορίας 26 υπέρ 33 κατά. Απορρίπτονται οι τρεις τροπολογίες. No. Yeah. So first eight is. Αν δεν κάνω λάθος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 221 ανάρχητη ψηφοφορία. Τέλος. 22 υπέρ 36 κατά. Απορρίπτεται. 219. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν ε, είχα ξαναδεί τέτοια διαφορά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 219 της καρτή Καταμάρα Λιωτάρ. Τέλος ψηφοφορίας, 25 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. 220 αν Φερέιρα, ποιος είναι υπέρ. Κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 220. Άρχεται ψηφοφορία. 25-32. Απορρίπτεται και αυτή. 222. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Άνια Βάισκερμπερ. 223. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επόμενη σελίδα. Δύο ταυτόσημες τροπολογίε οι 224 και 225. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνονται. Άλλες δύο ταυτόσιμες, οι 226 και 227. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 229 με προφορική τροπολογία του Φιέλνερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 229. Άρχεται ψηφοφορία. Χωρίς την προφορική τροπολογία όμως γιατί υπάρχει η αντίρρηση για αυτήν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 229 χωρίς την προφορική τροπολογία όμως. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ 36 κατά. Απορρίπτεται. 230 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Κάντε τη ζωή δύσκολη γιατί ακούγονται φυσαρίες. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. «48 υπέρ, 10 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 41 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίθηκε. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, 11 και 12 είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες 10, 11 και 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 25 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 13 της Γκιούλα Χέγγι. Οριακή θα είναι η διαφορά. 21 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο του της 14 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 24 υπέρ 32 κατά απορρίπτωται. Amendment. Επόμενη τροπολογία 15 να την ψηφίσουμε ή έχει καταπέσει. Ποιος είναι υπέρ τη 15, κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 15, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, 25 υπέρ, 33 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 16, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 17 πίπτη. 18 γκύλο χέτζι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 18 άρχεται ψηφοφορία The vote is closed. 28 in favor, 31 against. It has been rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ κατά ναι. αποχές απορρίπτεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ Against. κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 23 Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας 37 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. 24 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 24. Vote is closed. 37 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 25, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για καλό και για κακό για την τροπολογία 26 της Ούρσουλα Κρούπα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορίας. 21 υπέρ 34 κατά. Απορρίπτεται. 27 of Renata Zoma, who is in favor. Ε, Ζόμερ, 27 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 28 Ουρσούλα Κρούπα υπέρ. Κατά απόχέ Εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29 άρχεται ψηφοφορία τέλος 32 in favor, 25 against. It has been... Δηλαδή υπέρ 25 κατά εγκρίνεται. 30 της Ρενάτε Ζόμερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος καλύτερα. Για την 30. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλο vote 36 υπέρ 21 κατά αποχές. 31. Ποιος είναι υπέρ. κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 30. 2. The vote is closed. 21 in favor, 30 against. 21 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35, 36 και 37 ταυτόσιμες και η 38 το ίδιο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τέσσερις τροπολογίες 35, 36, 37 και 38 που είναι πανομοιότυπες ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία τέλος ψήφισαν 26 υπέρ 30 κατά απορρίπτονται απορρίπτονται είπα Ah. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It was. I. I can. Uh, I could read the numbers if if it would be necessary. It was. It... Συγγνώμη. Ήταν. Οι τέσσερις προηγούμενες, 26 υπέρ, 30 κατά και απορρίφθηκαν. 39, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 25 υπέρ 27 κατά. Απορρίπτεται. 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 και 41 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 42 της Χιλτρούδης Μπρέγερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 34 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 43. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 44. We are checking 44 and Ferreira's amendment and the vote. Αν Τέλος ψηφοφορίας. 27 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ιδια διαφορά, έλεγχος ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 45 της Άνε Φερέρα. Τέλος, 26 υπέρ 30 κατά, απορρίφθηκε και αυτή, 46 ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 και 48 ποιος είναι υπέρ. Και 49 47, 48 και 49. Τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ 47 έως 49. Καλά τα είπα στην αρχή. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίθηκαν αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος. 35 υπέρ 21 κατά. Εγκρίθηκαν. Η 50 καταπίπτει. 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 52 καταπίπτει. 54 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 54 Γκιούλα Χέτζη τέλος ψηφοφορίας 27 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται 53 Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ίδια διαφορά, γι' αυτό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, 25 υπέρ 31 κατά, απορρίπτεται. 4 πανομοιότυπες, 55, 56, 57 και 58. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 59, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος νομίζω ότι εγκρίθηκαν πάντως ε, η 59 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψήφισαν 35 υπέρ και 20 κατά όντως είχε εγκριθεί τέσσερις πανομοιότυπες 60, 61, 62 και 63 ποιος είναι υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τεσσερις τροπολογίες 60-63. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. 26 υπέρ 30 κατά απορρίπτονται. Δύο πανομοιότυπες 65 και 66. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Σαφώς έχει εγκριθεί 41 υπέρ, 14 κατά. Η επόμενη καταπίπτει 64 και τελευταία είναι 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 29 κατά. απορρίπτεται το σχέδιο έκθεσης. So 50 50 Okay. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Okay, we have so we, we have item 19, 17a now. Set Oh, okay. Light bulb. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση που μας έχει απομείνει είναι το 17α, έχει προσταθεί στην ημερήσια διάταξη και αφορά τη διαδικασία ε, επιτροπολογίας για τους λαμπτήρες φωτισμού. Just a second. Which has been circulated, prepare, prepare the draft. Σας έχει διανεμηθεί το κείμενο. Μία μόνο ψηφοφορία. Ο κύριος Τσίμπη θέλει το λόγο. Μπορούμε να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση του Μπογκούσου Αυσόνικ. Μόνο πέντε τροπολογίες έχει. Yeah, I'm, I'm sorry, I, I have no reason. Γιατί, γιατί να αλλάξει η σειρά των σημείων. Δεν υπάρχει λόγος. Μόνο μία ψηφοφορία θα γίνει της έκθεσης του κ. Κράμερ. Και υπάρχει συμφωνία, δεν διαφυσβητείται το θέμα. Ένα διαδικαστικό. Όπως είπα χθε, η ομάδα μου ζητά ονομαστική ψηφοφορία. Okay, Καλώς. Οι πράσινοι έχουν 17 μέλη. Πρέπει να σηκωθείτε παρακαλώ για να δούμε αν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ονομαστική ψηφοφορία. Χρειάζονται 17 ευρωβουλευτές. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah, more yeah. than 17. More than yeah, yeah, we have, we have 17. More than... 17. Εντάξει, έχουμε 17 ευρωβουλευτές και παραπάνω μάλιστα. Οπότε η πρόταση είναι σαφής, δεν χρειάζεται καν να τη διαβάσουμε. Είμαι ο μόνος που δεν την έχω μπροστά μου. ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζει ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Εντάξει, αφαιρέθηκε ψηφό. Ψήφισαν όλοι. Τέλο ψηφοφορία. 14 υπέρ, 44 κατά. Σαφώς απορρίπτεται το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ. Now let me jump to item 19. Πάμε στο σημείο 19 τώρα. And I would like to ask Boguslav Sonic if it's possible. Boguslav, κύριε Boguslav Sonic, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. So prepare your voting list. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία με τη συμφωνία του εισηγητού. The vote with amendments of Trapologia 3, Schlitter. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 5, τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. Το σχέδιο της γνωμοδότης όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας 43 υπέρ, χωρίς καμία αρνητική ψήφο και αποχή. Συγχαρητήρια θερμά κύριε Μποκούσοφ Σόνικ. Dear please, just, just few seconds. Συνάδελφοι, λίγα λεπτά ακόμη. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν πολύ δύσκολη αυτή η ψηφοφορία. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της πρωινής ημερήσιας διάταξης. Μην ξεχνάτε όμως ότι ε, μας έχει μείνει μια ψηφοφορία για το απόγευμα να βάλαμε το σημείο 16 για να το ψηφίσουμε το απόγευμα, έκθεση Σνέλχαρτ. Σας καλώ λοιπόν στην απογευματινή συνεδρίαση που θα ξεκινήσει